Καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Καθίστε. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση για τη συγκρότηση του Σώματος Επιτροπής ανάπτυξη. σύμφωνα με τη διάταξη 41 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου. Θα αναλάβω να διευθύνω την συνεδρίαση μέχρι του κληγή πρόεδρος της Επιτροπής μας. Να χαιρετήσω τους φίλους που επανεξελέγησαν, με τους οποίους έχουμε επί τόσα χρόνια συνεργαστεί. Που εργάστηκαν για την Επιτροπή για την προηγούμενη θητεία και επίσης σε θερμότατα καλωσορίσματα στους νέους συναδέλφους, εκείνους που ήρθαν στην Επιτροπή για πρώτη φορά. Πολύ ενδιαφέρουσα Επιτροπή ικανοποιεί πάρα πολύ κάποιον να ανταμείβει τη δουλειά του γιατί μπορεί να βελτιώσει, να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων που καμιά φορά συνέλακε του κόσμο που χωρί τη βοήθειά μα ίσω να μην ήταν καν στην ζωή ή δεν θα κάνει φαΐ να φάνε. Οπότε δεν μπορεί παρά να νιώσει κανεί ικανοποίηση ε, όταν εργάζεται εδώ σαν άνθρωπος και οπότε ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συγκυρία για όλους μας εδώ. Τέλο δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μα, οπότε χτίζει ο χρόνο να αρχίσουμε ευθύ αμέσω. Κυρίω την έναρξη τη ε, ε συνεδρίαση και όπω γνωρίζετε, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να συνηθούμε σε σώμα εκλέγοντα τον ε, πρόεδρο και το προεδρείο και τέσσερι δηλαδή αντιπρόεδρου σύμφωνα με την παράγωγη 204 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Πρώτον, θα εκλέξουμε τον την πρόεδρο κατόπιν στου τέσσερι. Αντιπρόεδρος. Από τις πολιτικές ομάδες έχω ε, λάβει τον νόματα των ανεπληρωτών οι οποίοι θα ε, ψηφίσουν και στον Δεμέρα για τον κύριο Μπεκιθερίλ, για το ΕΛΚ του Σκόζου, για τον κύριο Σόπλιν, για το ΕΛΚ επίσης, ο κύριος Χέις, για τον κύριο Στίερ, για το ΕΛΚ και ο φίλος Ρούμπιχ, αντί του κυρίου Πρέντα επίσης του ΕΛΚ. Κυρία Τόι για την κυρία Μάκαβαν, για τους Δημοκράτες και από την Παπανίληνα Μάκαβαν. Καθυστέρησε γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με το τρένο της, το κύριο Στάρ, ελπίζουμε εγκαίρως να βρίσκεται εδώ. Και Φανραμπ για την Ανιλίτς, για τους Σοσιαλδημοκράτες, ο κύριος Πρίνσκι για τον κύριο Γκερέρο των Σοσιαλιστών, κύριος Μάνσκο για τον κύριο Σίλβα Περέιρα, των Σοσιαλδημοκρατών επίση, ο κύριο Λου και τον κύριο Κάσκι τη ECR, Λέζινγκ, για τον κύριο Χρυσογόνο τη ε, ΓΚΟΕ. Αν υπάρχει κάποια αλλαγή, παρακαλώ να μου υποδείξουν οι πολιτικέ ομάδε ποια είναι αυτή η αλλαγή που έγινε πριν να So, let's proceed to Λοιπόν, ας εκλέξουμε, ας εκλέξουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, η απαρτία που απαιτείται είναι 7. Θα, θα πρέπει να επιψηφίσουν, έχουμε πάνω από 7 σήμερα εδώ. Τώρα για την υποψηφιότητα ή τις υποψηφιότητες για την θέση του Πρόεδρου. Έχετε το λόγο. Από πλευρά των Δημοκρατών προτείνω την Λίνα Μακάβαν ως πρόεδρο. Είναι στην Ευρωβουλή πάνω από 15 χρόνια. Έχει την εμπειρία, της ικανότητε, το ώστε να προεδρεύσει μεγάλη επιτυχία. Έχει ασχοληθεί με πολλά θέματα, περιβάλλοντο, αλλαγή του κλίματος δίκαιο εμπόριο, ανάπτυξη ε, παιδεία στι αντισωμένε χώρε και έχει επιδείξει ικανότητα συνεργασία με όλου του τέργε του Κοινοβουλίου και αυτό πιστεύουμε θα το κάνει και πάλι από τη θέση τη Πρόεδρου. Ευχαριστούμε για την πρώτη σχολή τη κυρία Λίντα Μακαβάν. Κάποια άλλη πολιτική ομάδα έχει να κατεβάσει κάποια υποψηφιότητα. Όχι. συμφωνείτε από πλευρά και για λογαριασμό τη για την υποψηφιότητα. Ναι, κύριε Νόιζα. Έχω λάβει μια εξουσιοδότηση από την Λίντα, ακριβώ για την κατάσταση των τρένων τη και είπε ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα. Έχει συμπληρώσει την δήλωση οικονομικών συμφέροντων, είναι τακτικό μέλος και δέχεται την υποψηφιότητα για την θέση της Πρόεδρου. Μια που υπάρχει μόνο μία υποψήφιος για την θέση του Πρόεδρου, σας προτείνω να την εκλέξουμε διαβοής. Thank you, colleagues. Ευχαριστώ συνάδελφε. Επομένως, να κηρύσουμε ως πρόεδρο της ε, Επιτροπής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου διαβοή στην κυρία Μακρόν και θα τις διαβάσω και από πλευρά σας τα συγχαρητήρια όταν την συναντήσω. Τώρα θα έπρεπε να δώσω τη θέση μου σε εκείνη, δεν βρίσκεται εδώ, οπότε θα συνεχίσω για να εκλέξουμε τους αντιπρόεδρους. remind you of the names of the substitutes that να σας ε, υπενθυμίσω τα ονόματα των αναπληρωτών που θα συμμετάσχουν στην πληροφορία για τους ε, αντιπροέδρους. Νομίζω ότι επειδή το έκανα πριν δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνω και τώρα μάλλον. Οπότε προχωρούμε στην ψηφοφορία για τους αντιπροέδρους. Ξεκινούμε με τον πρώτο αντιπρόεδρο. Θα ήθελα να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Παρακαλώ. Κύριε Βέντε. Εντάξει. Θα ήθελα εκ μέρου του ΕΛΚ να προτείνω τον κύριο Μωρίς Πονγκά για τη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Ευχαριστώ. Μωρίς, συμφωνείς με την υποψηφιότητά σου. Ναι. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο υποψήφιο θα πρέπει να είναι τακτικό μέλος τη επιτροπή και να έχει συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Πληρούνται αυτέ οι προποθέσει. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα για την θέση του πρώτου αντιπροέδρου Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης. Επομένως, προτείνω να ε, εκλέξουμε τον κύριο Πόγκα διαβοή. Um, Ευχαριστώ. Συγγνώμη που, που καθυστέρησα. Για όσους δεν γνωρίζετε, ε, υπήρχαν προβλήματα ε, με το Eurostar σήμερα όλη μέρα, οπότε πάρα πολλοί ευρωβουλευτές από τη Βρετανία αυτή τη στιγμή εισραίουν στο κτίριο. Χαίρομαι πολύ που ε, προτάθηκα και εξελέγην πρόεδρος. Έχουμε σημαντικό έργο τα επόμενα χρόνια. Έχουμε την αναθεώρηση των στόχων για την ανάπτυξη. Το 2015 είναι έτος αγροτικής ανάπτυξης και Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε. Σήμερα όμως δεν είναι ε, η συνεδρίαση για να εκφωνούμε λόγους. Θα συνεχίσουμε με την επόμενη ψηφοφορία και ζητώ αυτή τη στιγμή να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τη θέση του δεύτερου του Προέδρου της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, οι υποψηφιότητες. Yes, thank, you, Mr. Ναι, κύριε θα ήθελα από τη σειρά μου να σας συγχαρώ κυρία Πρόεδρε που αναλάβατε καθήκοντα Προέδρου της ε, Επιτροπής μας και την υποψηφιότητα του Παύλου Βαρούνεν ε, για τη θέση του Αντιπροέδρου από πλευράς της Άλντε. Ευχαριστώ κύριε Γκέρεν, άλλη πολιτική ομάδα. Έχει άλλο υποψήφιο. Κύριε Βερένεν, είστε εκεί. Δέχεστε την υποψηφιότητα. Δέχομαι. Να σας υπενθυμίσω ότι σαν υποψήφιος πρέπει να είσαστε πλήρες μέλος της Επιτροπής και να έχετε δεόντως συμπληρώσει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Ε, πληρούνται αυτά τα κριτήρια. Απάντηση. Μάλιστα κυρία. Καλώς λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Εν αυτή η περιπτώση συνάδελφοι έχουμε μόνο έναν υποψήφιο για θέση δευτέρου αντιπροέδρου της Επιτροπής, οπότε προτείνω να εκλεγεί ο κ. Βερέινεν διαβοής. well... Και παρακαλώ να έρθετε να πάρετε τη θέση σας στο Προεδρείο της Επιτροπής. Πάμε λοιπόν για θέση αντιπροέδρου, του τρίτου αντιπροέδρου, της τρίτης αντιπροέδρου της Επιτροπής. Εν ονόμα της ΓΚΟΕ, NGL, υποψηφιότητα για θέση του τρίτης αντιπροέδρου στον κύριο Κώστα Χρυσογόνο. Με την, έχει την απόλυτη υποστήριξη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες από άλλη πολιτική ομάδα. Όχι. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσόγονος απουσιάζει, αλλά δέχτηκε την υποψηφιότητά του γραπτός και είπε ότι είναι πλήρες μέλος αυτής της Επιτροπής και έχει συμπληρώσει την δήλωση του περί οικονομικών συμφερόντων. Άρα μπορούμε να εγκρίνουμε τη θέση, το διορισμό του θέση του Αντιπροέδρου διαβοή. Μπορεί να απουσιάζει, αλλά μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία εκλογής του διαβοή. Τελευταία εκλογή για Αντιπρόεδρο, τέταρτου Αντιπρόεδρου τη Επιτροπής. Υποψηφιότητες παρακαλώ. Κύριε Λούκα, για την ομάδα ECR. Τον κύριο Νάτζ Δίβα προτείνω. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα από άλλη πολιτική ομάδα. Ο κύριος Δίβα. Α, εκεί είσαστε. Κύριε Ντίβα, δεχόσαστε την υποψηφιότητα. Ναι, κυρία Πρόεδρε. Πληρούνται οι προποθέσει, είσαστε πλήρε μέλο, συμπληρώσατε τη δήλωσή σα περί οικονομικών συμφερόντων. Ναι, απαντάει ο κύριο Ντίβα. Ναι, ναι. Οπότε έχουμε έναν υποψήφιο μόνο Λοιπόν, ξανά διαβοή σας καλωσορίσουμε τον κύριο Ντέβα. Και τον ευχαριστώ που ξεκίνησε τη διαδικασία, ήταν πρόεδρος της συνεδρίασης. Δύο θητείες ήταν, τρεις θητείες ήταν μέσα Επιτροπής. Μάλιστα, τον θυμάμαι προηγούμενες θητείες. Με τα χαρά σας βλέπω εδώ. Οπότε ολοκληρώνεται η εκλογή των αντιπρόεδρων. Τρίτο σημείο της σα διάταξη είναι το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων για το υπόλοιπο 2014. Να πω στους νέους ε, συναδέλφους ότι θα δείτε ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 22 Ιουλίου στις 3 δεν έχω ακόμα αίθουσα να πω στα νέα μέλη επίση ότι καμιά φορά πρέπει να προσθέσουμε έκτακτε συνεδριάσει και αυτέ μπορεί να είναι Στρασβούργο, Δευτέρα, απόγευμα, Πέμπτη πρωί. Θα σα ειδοποιεί εγκαίρω η γραμματεία για τυχόν πρόσθετε συνεδριάσει. Για την ώρα αυτά έχουμε προγραμματίσει για φέτο και αργότερα το φθινόπωρο θα εγκριθεί και το πρόγραμμα των συνεδριάσεων του 2015. Συμφωνείτε λοιπόν με τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων μας του 2014. Ναι, δεν υπάρχουν προβλήματα. Καλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεκτές ημερομηνίε και συμπληρώστε στα... στο πρόγραμμά σας. 22 Ιουλίου είναι η συνεδρίαση, σας το είπα και αυτό. Εξετάστε τα εγγραφά σας, νέοι συνάδελφοι. Σας ειδοποιούμε, σας στέλνουμε και έγγραφα για τις συνεδριάσεις. Υπάρχουν τα έγγραφα εκ των προτέρων στο διαδίκτυο, βρίσκετε τα έγγραφα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, έχετε στη διάθεσή σας τη γραμματεία και η γραμματεία θα σας παρουσιαστεί και θα σας συστηθούν τα μέλη της γραμματείας με την πάρα των συνεδριάσεων. Μην διστάζετε να θέσετε ερωτήματα. Όταν κανείς έρχεται για πρώτη φορά, πολύ συχνά τα πράγματα φαίνονται δύσκολα. Λέει κανεί δεν ξέρω πώ λειτουργούν αυτά. Είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε κόσμο στη γραμματεία που μπορεί να σα βοηθήσει και στι πολιτικέ ομάδε σα. Επόμενη συνεδρίαση λοιπόν. 22 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μα. Ευχαριστώ πολύ που ανεχθήκατε την καθυστέρησή μου. Όπω σα είπα όμω, θα έχουμε χρόνο στην επόμενη συνεδρίαση ελπίζοντα, ώστε να παρουσιαστούν οι διάφοροι συνάδελφοι, να συσταθούν και να ξεκινήσουμε τι εργασίε μα για την επόμενη πενταετία. Ευχαριστώ πολύ.